η οποία αποτελεί το αντικείμενο αίτησης άρσης της ε, βουλευτικής ασυλίας διότι έχει εμπλακεί σε κάποια δίκη ε, εναντίον της στην Βουδαπέστη. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει υποβάλει κάποιες υποψηφιότητες για τις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές. Όλα αυτά θα καταχωρηθούν εις τα πρακτικά, εάν δεν υπάρχει παρατήρηση ή ένσταση μέχρι την μοστική ε, έγκριση των πρακτικών, οπότε και υπ' αυτή την επιφύλαξη οι προτάσεις του ΕΛΚ θα εγκριθούν. Od 1 2010